E, tego protokołu. Bardzo proszę, pan poseł Golnisz. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω δυνάμει του άρθρου 172 στο σημείο 5.2 των πρακτικών του Σεπτεμβρίου και θα εστιάσω την παρέμβασή σου δυνάμει του άρθρου 145. Κύριε Πρόεδρε, ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα ψηφίστηκε που καταδικάζει τη γαλλική κυβέρνηση για την πολιτική που, ε, απέλασης που εφαρμόζει για τους νομάδες ε, και τους Ρώμα. Αυτή η ψηφοφορία παραδόξως παρόλη τη σημασία της δεν υποβλήθηκε στις ομάδες που ε, ώστε να, μπορέσουν, να μπορέσει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Παρόλο που εγώ και οι πολιτικοί φίλοι μου ανήκαμε στη μειοψηφία <clears throat> που καταψήφισε αυτό το ψήφισμα που καταδικάζει τη γαλλική κυβέρνηση, αποτελέσαμε τη μειοψηφία των 240 βουλευτών που ψήφισαν κατά ορισμένοι συνάδελφοι, ο κύριος Ρομπιέ Ροντί και η κυρία Βερονίκ Μαντιό ειδικότερα συγκεκριμένα, ισχυρίστηκαν ότι ψηφίσαμε το ψήφισμα που καταδίκασε τη γαλλική κυβέρνηση κάτι που θα μπορούσε να είναι ένα λάθος εξελίχθηκε σε κρατικό ψεύδος όταν το επανέλαβε ο υφυπουργό για ο κύριος Πιέρ Λουλούς και ο κύριος Ζων Φρανσουά Κοπέ η παρέμβασή μου στη συζήτηση, οι εξηγήσει ψήφου που έδωσα, η προσπάθειά μου να αντισταθώ σε αυτά που ήθελε να κάνει ο κύριο Βόμποντα ήταν απόλυτα σαφή. Γιατί δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία. Αντίθετα με αυτό που σε εδώ, είναι παρέμβαση, σαφώς παρέμβαση του ΕΛΚ, έγινε μια προσπάθεια, έγινε μια προσπάθεια να κατηγορηθεί να μας κατηγορήσουν οι αντίπαλοι μας. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας κυρίες και κύριοι. Αν κατάλαβα καλά, αυτή ήταν μια παρατήρηση σχετική με τα πρακτικά και τις προσωπικές δηλώσεις. Ήταν μια αναφορά στις ε, παρεμβάσεις σας τις προηγούμενες. Έχετε κάποια άλλα σχόλια να κάνετε για τα πρακτικά της 9ης με 13 Σεπτεμβρίου. Γίνονται δεκτά. Κάποιες επιπλέον πληροφορίες